Λοιπόν, σας ε, καλώ αύριο να υπερψηφίσετε αυτή τη συμβαστική λύση έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έκλεισε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Τώρα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε ό,τι αφορά τη θέση του Αντιπροέδρου που χείρεψε, έχω τις ε, εξής ε, υποψηφιότητες από το ΕΛΚ, Λάσλο Τόκες. Η εκλογή θα γίνει αύριο, 3η 15 Ιουνίου 2010, στις 12 η ώρα του μεσημέρι. Και τώρα, με βάση την ε, ημερήσια διάταξη, έχουμε την έκθεση Λάτφορτ σχετικά με τα δικαιώματα σε διερμηνία και μετάφραση στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λάτφορτ, που είναι η συγγήτρια. Έχετε το λόγο. It's been recognized by most... Εδώ και δέκα χρόνια περίπου έχουμε να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει για να ενδυναμώσει τα δικαιώματα των ε, κατηγορουμένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δίκαιη δίκη. Ε, θα πρέπει η εισαγγελία και οι αστυνομικέ αρχές να συνεργαστούν πολύ πιο στενά από ό,τι για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Σύλληψης. Εδώ πέρα ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν απόπειρε για να εξασφαλιστούν τα δικονομικά δικαιώματα, κάτι που θέλουν οι ευρωβουλευτές. Το 2007 έγινε μια προσπάθεια. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χαίρομαι που είναι παρούσα η κυρία Ρέντινγκ για αυτή τη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υποστήριξη της Σουηδικής Προεδρίας ε, ανανέωσε υπό τη μορφή ενός οδικού χάρτη την προσπάθεια αυτή. Ε, και φτάσαμε σε αυτήν την οδηγία. Αν είσαστε ύποπτος, αν έχετε συλληφθεί ή αν περνάτε από δίκη, αν δεν καταλαβαίνετε τη γλώσσα της χώρας, έχετε το δικαίωμα ε, σε διερμηνία και μετάφραση υπό κάποιους όρους ε, κατά τις από την αστυνομία, για τις ακροάσεις, τις συναντήσεις με τον δικηγόρο σας κτλ. Γενικά, θα πρέπει να είστε στην ίδια θέση όπως και οι γηγενείς. Η βάση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών ε, στις ποινικέ ε, δίκες είναι η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων των δικαστηρίων σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν είναι λογικό όμω να υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη απλά και μόνο. Θα πρέπει να κερδιθεί ε, με το σεβασμό των προτύπων από όλε ε, τις χώρες κάποιων προτύπων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι δεν έχουν ε, περάσει δίκη. όπως παραδείγματο χάρη ο Γκάρι Μαν, ο οποίος συνελήφθη στην Πορτογαλία με βάση το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ο κύριος Μαν δεν ήξερε γιατί τον κατηγορούσε παρά μόνο όταν τον, τον καταδίκασαν. Όταν επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, του έστειλαν απλώ ένα γράμμα και του είπαν μην ξαναπατήσει ε, στην ε, Πορτογαλία. Ε, ο άνθρωπο αυτό ήταν ένα απλό κομμωτή, δεν γνώριζε την, ε, την πορτογαλική γλώσσα. Ε, Επίσης ο Άντριου Σίμιου σε μια υπόθεση δίκη στην Ελλάδα επίσης δεν γνώριζε ελληνικά. Έχουμε το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ε, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται ε, και θα πρέπει να ε, εξασφαλιστούν και κάποια άλλα δικαιώματα πέρα από τα ελάχιστα πρότυπα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουμε την πλήρη, τον πλήρη σεβασμό των στάνταρ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και μάλιστα όχι απλώς να τα σεβαστούμε αλλά να τα αυξήσουμε. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί καλά τις νέες του εξουσίες με βάση τη Λισαβόνα. Πολεμήσαμε μαζί με την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ, τη συγχαίρω γι' αυτό, για να αυξήσουμε τα πρότυπα ε, σε ό,τι αφορά τη διερμηνία, την επικοινωνία μεταξύ του κατηγορουμένου και του ε, δικηγόρου του σε όλες τις φάσεις της ε, δίκης. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένδικα μέσα, έχει το δικαίωμα στη μετάφραση και έχει το δικαίωμα να για την ποιότητα. Επίσης, όλα τα έγγραφα θα πρέπει, τα ουσιαστικά έγγραφα θα πρέπει να μεταφράζονται. Ο ύποπτο δεν θα πρέπει να παρατείται από το δικαίωμα της μετάφρασης χωρίς ε, ε, συζήτηση. Χρειαζόμαστε το πρόγραμμα του οδικού χάρτη, ούτως ώστε ε, να λειτουργήσουν καλύτερα τα δικαιώματα, ε, η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων της υπεράσπισης δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πιο μαλακοί απέναντι στους εγκληματίες. Αντίθετα, καλές αποφάσεις σημαίνει ότι πιάνουμε περισσότερους εγκληματίες. Ε, και η μείωση των ε, δαπανών ε, δεν νομίζω ότι οδηγεί σε καλές και ποιοτικέ δίκες γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε περισσότερε Ε, Ευθυνή δικαιοσύνη σημαίνει κακή δικαιοσύνη. Ε, μαζί με την Ισπανική Προεδρία είχαμε καλές διαπραγματεύσεις καθώς και με την Επιτροπή όπως σας είπα όταν ε, ε, κλείσω στη δευτερολογία μου, λέτε, θα σας μιλήσω για τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Και τώρα η Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, σωστά. Διαδικαστικά πρέπει κανείς ε, να ε, είναι προφυλαγμένος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα επόμενα έτη. Χρειάζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα ε, των κατηγορουμένων σε ποινικέ διαδικασίες και πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών των διαφόρων κρατών διότι χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ε, αμοιβαία αναγνώριση. Θα πρέπει και οι εισαγγελείς και οι δικαστές ε, να ε, μπορούν να επαναπαυθούν ότι οπουδήποτε υπάρξει μία δίκη στην Ευρώπη θα ισχύσουν τα ίδια μέτρα και σταθμά και θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικαιώματα τα οποία θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο δικαστικό σύστημα και γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω θερμά τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι δύο συνομοθέτες και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τη Βαρόνη Λατφόρτ και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την εξαιρετική εργασία που έκαναν σε αυτό το τομέα. Η, Επιτροπή θεωρεί ότι πολλές από τις συμβιβαστικές λύσεις ξεκινούν και εμπνέονται από την πρότασή μας για την πρόοδο του 2010. Δηλαδή αυτό το οποίο ε, επιζητούσαμε να επιτύχουμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και ε, ε, μην είναι υποδέστερα από το κεκτημένο <clears throat> για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη πρέπει να υπάρξουν ελάχιστες προδιαγραφές, να υπάρχει ενιαία ερμηνεία κατά την δικαστική διαδικασία και η μετάφραση των εγγράφων να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μία δίκαια δίκη. Συμφωνώ πλήρως με την εισηγήτρια. Η φθηνή δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη και οδηγεί σε μεγαλύτερα έξοδα στο τέλος και δεν υπάρχει και καμία εμπιστοσύνη ούτε από πλευράς δικαστών ούτε από πλευράς πολιτών. Γι' αυτό και χαίρομαι ότι μπόρεσε να υπάρξει μια ταχεία υιοθέτηση αυτής της οδηγίας και είναι ένα βασικό στοιχείο του χάρτη πορείας κατά τρόπον ώστε όλοι οι πολίτες να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για ένα θέμα προτεραιότητος. Υπάρχει μόνο ένα σημείο στο οποίο διαφωνώ κυρία Πρόεδρε. Και αυτό είναι η αίτηση από ορισμένε χώρες οι οποίες ε, ζητούν να ε, ε, ε, καθυστερήσει κατά 36 μήνες η εφαρμογή. Θεωρούμε ότι τρία χρόνια επιπλέον είναι περιτά και λανθασμένα διότι δεν θεωρούμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ισχύσει σωστά η διαδικασία και εντωμεταξύ θα υπάρξει και νέα νομοθεσία. Ε, αυτό ούτως ή άλλως ήταν γνωστό εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε ε, έχω κάνει την παρατήρησή μου αλλά συμβιβαστικά θα σας πω ότι δέχομαι μία λύση και αυτό που σας λέω είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον ε, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό δεν θα αποτελέσει ένα προηγούμενο για μελλοντικά μέτρα του χάρτη πορείας και το τονίζω τρεις φορές. Ναι μεν στην περίπτωση αυτή θα το δεχτούμε αλλά τελευταία φορά και όχι περαιτέρω. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει για να ενισχύσει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών να εφαρμόσουν εγκαίρως και σωστά την απόφαση σύμφωνα με την συνθήκη της Λισαβόνας και ε, τα συμπεφωνημένα. Ξέρετε βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προετοιμάζει τα μέτρα του επομένου χάρτη πορείας και σύντομα θα σας δώσω την πρόταση για το δικαίωμα για πληροφόρηση εντός των επομένων εβδομάδων άρα αυτό που ξεκινήσαμε σήμερα θα προχωρήσει γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε και τώρα στρέφομαι εις τους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Καταρχήν η κυρία Αντωνέσκου εκ μέρους του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια κυρία Λάτφορντ για τη δουλειά της αλλά και για τη συνεργασία που είχε με τους άλλους εισηγητές. Τα κοινά πρότυπα είναι απαραίτητα για να υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη στα νομικά συστήματα των κρατών μελών. Τα δικαιώματα δίκαιη δίκη των υπόπτων ή κατηγορουμένων είναι ένα θεμελιώδε δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίες. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν αξιοπρεπή πρότυπα υπεράσπισης θα υπάρχει ανισορροπία μεταξύ ε, των ε, μέσων που χρησιμοποιεί ο εισηγητή και των ε, μέσων που έχουν στη διάθεσή του οι ε, υπόπτη κατηγορούμενοι. Η ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μακρά συνεχιζόμενη διαδικασία. Το Νοέμβριο του 2000 έγιναν τα πρώτα βήματα και το Συμβούλιο, ε, με βάση τα συμπεράσματα του Τάμπερε, υιοθέτησε ένα εκτελεστικό πρόγραμμα για την αμοιβαία αναγνώριση σε θέματα ποινικά. Είχαμε την πρόταση τη Κομισιόν για μια απόφαση πλαίσιο το 2004. Δεν κατέστησε δυνατή επίτευξη συμφωνία και το 2007 τον Ιούνιο ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις. Επίσης το 2009 είχαμε τον οδικό χάρτη της Σουηδική Προεδρίας που πρότεινε μια ε, σταδιακή προσέγγιση στα δικονομικά δικαιώματα. Η πρόταση της Κομισιόν τον Ιούλιο του 2009 και τον Δεκέμβριο του 2010 και το Δεκέμβριο του 9 μάλλον, και έπειτα έχουμε αυτή την πρόταση για τα 13 κρατημέλη. Μετά από 7 χρόνια λοιπόν φτάνουμε να εγκρίνουμε τα πρώτα μέτρα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη και μιλώ για αυτή την οδηγία για τα δικαιώματα στη μετάφραση και τη διερμηνία. Είμαι πολύ ικανοποιημένη με τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μετά τι διαπραγματεύσει μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ένα κείμενο το οποίο συνιστά σημαντική βελτίωση στην αρχική πρόταση. Ελπίζω η περίοδος εφαρμογής των τριών ετών να μην αποτελέσει προηγούμενο για τα προσεχή μέτρα στο πλαίσιο του οδικού χάρτη και ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να εφαρμόσουν συνεκτικά και ταχαίως όλες τις διατάξεις οδηγίας. Η κυρία Ρομέρο Λόπεθ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εμένα με ικανοποιεί που βλέπω ότι οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται και θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Λάτφορτ όλους ιδιαιτέρως και για την συνεργασία με την οποία είχαμε όλοι οι σκιώδες τις μαζί της. Είναι η πρώτη περίοδος συναπόφασης, ε, περίπτωση συναπόφασης που είχαμε σημαντική συμβολή ως ε, κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι μια Αγγλίδα Ευρωβουλευτής είναι αυτή που ανέλαβε ε, τη σύνταξη της έκθεσης για αυτή για αυτό το θέμα. Χρησιμοποίησε λοιπόν ε, το προνόμιο που του έχει χορηγηθεί από την ε, Συνθήκη της Λαβώνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υποβάλει αυτή την πρωτοβουλία που υπέβαινε τρία μέλη. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση του 2004 για τα δικονομικά δικαιώματα, έχουμε μια μερική απεμπλοκή του στον οδικό χάρτη που παρουσίασε η Σουηδική Προεδρία. Άρα είχε ανοίξει δύο δρόμος, ο οποίος όμως διεκόπη όταν εξελέγει νέα επιτροπή. Στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει την πρώτη πρόταση οδηγίας την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις τροπολογίες του έλαβε υπόψη τις ε, εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να ένα παράδειγμα καλής θεσμικής συνεργασίας για να μην χάνεται χρόνος και για να υπάρξει ε, μια ευελιξία και γρήγορη δεκπεραίωση αυτών των δικονομικών διαδικασιών. Υπήρξε λοιπόν αυτή η ταχύτητα στη δεκπεραίωση και τώρα όπως είπε και η Επίτροπος είναι καιρό στα άλλα δικαιώματα, ο χάρτης των δικαιωμάτων ε, που είναι η δεύτερη δέσμη στο πλαίσιο των δικονομικών αυτών δικαιωμάτων είναι το δεύτερο κομμάτι και επίσης υπάρχει και κάτι ακόμη γιατί δεν θα είχε κανένα νόημα να υπάρξει καθυστέρηση με αυτό το πακέτο και να μην ολοκληρώσουμε μέσα σε εύλογα χρονικά πλαίσια ε, η ελευθερία δικαιοσύνη ασφάλεια. Δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί αν δεν βάλουμε τα θεμέλια των, των δικονομικών αυτών εγγύσεων για να έχουμε μια ελεύθερη ασφαλή ε, δίκαια, ε, ένα δίκαιο χώρο στον οποίο θα ζούμε. Πώς θα γίνει αυτό αν δεν υπάρχουν αυτέ οι δικονομικέ εγγύσει, οι ελάχιστε αυτές εγγύσει στα κράτη-μέλη για υπόψη και κατηγορουμένους. Τι θα σημαίνει λοιπόν αυτή η Ευρώπη που θέλουμε να οικοδομήσουμε και όπω είπαν και άλλοι συγητές, οι τρομοκρατικέ απειλέ, το οργανωμένο έγκλημα μα υποχρεώνουν να ενισχύσουμε του μηχανισμού ασφαλεία. Γνωρίζουμε όμω, εξού και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, γνωρίζουμε όμω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταφέρουμε να. Μάλλον, αν δεν καταφέρουμε να έχουμε την Ευρώπη τη ελευθερία, ασφάλεια δικαιοσύνη, δεν θα έχουμε αυτό το ασφαλέ μέλλον που όλοι ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ. Και τώρα, μία ερώτηση από, την, από τους φιλελεύθερους. Κυρία Ρομέρο Λόπες. Κυρία Ρομέρο Λόπες. Υπάρχει μια ερωτηση απο την τους φιλελευθερους κυρια ρομερο λοπες κυρια ρομερο λοπες υπαρχει μια ερωτηση για σας. Από Από το ΔΙΚΑ... τον γκόμι Ντάρμουθ. Έχει 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Οι πολίτες σε χώρες που έχουν πολύ ψηλότερα πρότυπα ατομικών δικαιωμάτων, παραδείγματο χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπόκεινται σε χαμηλότερα, ε, ε, στο χαμηλότερο επίπεδο δικονομικών δικαιωμάτων που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη και με βάση τις ευρωπαϊκές ε, οδηγίες που ισχύουν. Το ξέρετε εσείς αυτό. Τι έχετε να απαντήσετε. Eh, Ή, κοιτάξτε, μάλλον ε, ερώτηση ουσιαστικά αναφέρεται σε αυτά τα ελάχιστα πρότυπα τα οποία εμείς ζητούμε ε, για τα διάφορα κράτη-μέλη ε, και θέτει κάπω υποαμφισβήτηση όλο αυτό. Εγώ θεωρώ ότι κάθε χώρα μπορεί να θεσπίσει τα δικά της ε, πρότυπα, αλλά η πρόθεση κάθε χώρα νομίζω είναι να οικοδομήσει μια Ευρώπη που θα είναι ευπρόσδεκτη, φιλόξενη και όπου θα έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα και κάποιε ελάχιστε εγγύσεις για όλου. Ξέρουμε την ιστορική παράδοση της χώρας σας αλλά και πολλών άλλων ε, χωρών που αποτελούν αυτή την Ευρώπη γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι θα αυξηθούν όλο και περισσότερα αυτά τα πρότυπα. Πάμε τώρα στους ε, ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Κυρία Τάιν, από την ομάδα των Φιλελευθέρων, για ένα λεπτό. Sehr geehrte Αξιότιμες κυρίες και κύριοι ε, για να μπορέσουμε να πατάξουμε με καλύτερο τρόπο την εγκληματικότητα στην Ευρώπη χρειάζεται ε, στενότερη συνεργασία και αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως. Υπάρχουν όμως και τα δικαιώματα των κατηγορουμένων τα οποία δεν έχουν ε, προστατευθεί και γι' αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή να συμφωνήσει ομόφωνα το Συμβούλιο για να προχωρήσει η αμοιβαία αναγνώριση και αυτό έχει αποτύχει. Θα πρέπει λοιπόν να προφυλαχθούν τα δικαιώματα των ε, πολιτών ε, για τις ε, ποινικέ διαδικασίες και γι' αυτό ζητούμε στο μέλλον όλοι οι πολίτες να έχουν δικαίωμα σε διερμηνία και γραπτή μετάφραση όταν κατηγορούνται σε ένα κράτος το του οποίου δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Δηλαδή ε, θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός καλύτερος για να καλύπτονται τα δικαιώματα των πολιτών, όλοι να έχουν μία ε, δίκαια αντιμετώπιση ε, και ευχαριστώ. Κυρία Χάουτα, από τους Πράσινους για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ερώτημα το οποίο τέθηκε προς την κυρία Ρομέρο Λόπες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ακριβώς γι' αυτό δουλεύουμε, για να υπάρξουν ελάχιστες προδιαγραφές για τα δικονομικά δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορούμε να εμπιστευόμαστε α, το τι γίνεται σε τι άλλο, αυτό που, γίνεται, που συμβαίνει σε άλλα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη θαυμάσια δουλειά, που έγινε ε, και τη θαυμάσια συνεργασία με τους σκιώδει εισηγητέ. Να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια οδηγία τώρα που θα εγγυάται σε όλου τη δυνατότητα να καταλάβουν ε, τι τους λένε και να μιλήσουν και να τους καταλαβαίνουν ε, κατά τις ποινικές διαδικασίες. Αυτή είναι προϋπόθεση για την καλή διεξαγωγή των δικών. Ευχαριστώ τον εισηγητή που προσπάθησε να βρει λύσει, να υπερβληθούν οι δυσκολίες που υπάρχουν σε διάφορα κράτη-μέλη λόγω των διαφορών ε, στις αρχές δικαίου. Φυσικά η θέση σε ισχύ και οι 36 μήνε προθεσμίας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι πρέπει να δεχτούμε αυτό το αποτέλεσμα γιατί είναι κάτι που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής δεν είναι εδώ. Γι' αυτό θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ντεμπρούν από την ΚΟΕ για 1,5 λεπτό. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ζήτημα ε, το οποίο δυστυχώς ε, αντιλήφθηκα πολύ αργά και δεν μπόρεσα να, να καταθέσω ε, τροπολογία θα ήθελα να σχολιάσω. Χαιρετίζουμε την αναφορά στο δικαίωμα μετάφρασης, διερμηνία, στο να μπορεί να μιλεί ο ή κατηγορούμενος στη μετρική του γλώσσα, στο 10 γ συγκεκριμένα του συμπεφωνημένου κειμένου. Υπάρχει ωστόσο ένα κίνδυνο. αυτός, αυτή η έκφραση που λέει η μητρική γλώσσα ή οποιαδήποτε γλώσσα κατανοεί, εκεί μπορεί να οδηγήσει αυτό σε περιορισμό ε, των γλωσσών. Δηλαδή να αναγκαστεί ο ύποπτο ε, κατηγορό να χρησιμοποιήσει γλώσσα που δεν είναι ε, γλώσσα τη επιλογή του ή τη επιλογή τη. Και βέβαια όταν έχουμε να κάνουμε πολύπλοκα δικονομικά ζητήματα καταλαβαίνετε τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Θα μπορούσε η Επίτροπος να υποσχεθεί ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο και ότι και οι μειονοτικές γλώσσες θα ληφθούν υπόψη Οι τροπολογίε μα που υποστηρίζονται και από μέλη άλλων πολιτικών ομάδων αναφέρονται σε ευρωπαϊκά διεθνή ε, μέσα και πράξεις ε, που προασπίζουν τα δικαιώματα και τις ε, μειονοτικές γλώσσες. Και αναφερόμαστε συγκεκριμένα ε, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ευρωπαίων Δικαιωμάτων που μιλά για αυτά τα δικαιώματα. Ελπίζω το θέμα των γλωσσών να διευκρινιστεί εγκαίρω. William Κύριε, κυρία Πρόεδρε, η οδηγία αυτή είναι στο πλαίσιο μια σειρά οδηγιών που έχει αποτέλεσμα κάθε πολίτη και κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου να μπορεί να μπει ε, στα κάτεργα σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αν αυτή η χώρα τώρα είναι η Πορτογαλία, στην περίπτωση του Γκάρι Μαν, η Ουγγαρία, σε περίπτωση ε, δύο κατοίκων ε, της από το Southwest, αυτό δεν αλλάζει το ότι δεν υπάρχει ίδια νομική προστασία για τους πολίτες όπως αυτοί που θα είχαν στον Ηνωμένο Βασίλειο παρά των αυταπατών που μπορεί κανείς να έχει σε αυτό το κοινοβούλιο. Επομένω, η αυτή οδική για τη μετάφραση είναι ένα φιλοσικής Προσπαθεί να κολλήσει ένα χαντζαπλάστ ε, στο σημείο που σχεδόν ε, βλέπουμε να έχουν ακροτηριαστεί οι πολύ σκληρά κατακτημένες ελευθερίες Βρετανίας από το χέρι του Ευρωπαϊκού ε, Εντάλματος Σύλληψης. Είναι λοιπόν λάθος η οδηγία αυτή. Η απόφαση ουσιαστικά για τη μετάφραση έγκυται σε μεγάλο βαθμό στον Γενικό Εισαγγελέα και επίσης στην κατηγορούσα στο δημόσιο κατήγορο. Και επίση υπάρχει χρόνια και μεγάλη έλλειψη μεταφραστών και διερμηνέων. Και γιατί απορροφώνται πολλοί από αυτού από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διακεκριμένη συνάδελφό μου Βαρόνι Λάτφορτ πολλές φορές λέει ότι είναι ε, υπέρμαχο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Την ε, ζητώ, τη ζητώ λοιπόν για μια φορά να βάλει κατά μέρο την ψύχωση που έχει για την Ομοσπονδιακή Ευρώπη και να έρθει στη δική μα να προσετεριστεί ε, τα στρατόπεδό μα για την κατάσταση του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ και περνάμε τώρα στου ομονωμένου ομιλητέ. Πρώτα απ' όλα στον κύριο Μπούσιτλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η πρόταση είναι εξαιρετική και πρέπει να στηριχθεί διότι <clears throat> δίνει περισσότερα δικαιώματα εις ε, τους πολίτες. Το ΕΡΚ θα υπερψηφίσει αυτό τον κανονισμό αλλά όχι τις ε, τροπολογίες γιατί θα διαταράξουμε την ισορροπία που επετεύχθη. Στα σχόλιά μου θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, αφήσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποβολή της προτάσεως αυτής. Διότι δεν έχουμε μία πρόταση, έχουμε δύο προτάσεις. Τον ε, Δεκέμβριο ε, υπήρξε η πρόταση του Συμβουλίου των Υπουργών και το Μάρτιο η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του ιδίου θέματος. Με αυτόν τον τρόπο ε, έρχομαι στην ερώτησή μου. Δηλαδή ε, ποιο κείμενο είναι αυτό το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσει σαν βάση των συζητήσεών μας στο Κοινοβούλιο και δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι κάτι που θα συνεχίσει να προκύπτει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, την πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη μας είπε ότι θέλει να διατυπώσει μία νέα πρόταση. Και τώρα το Συμβούλιο μας λέει ότι πρέπει να δεχθούμε αυτό το, αυτή την πρόταση ενώ η Επιτροπή μας ζητά να μην την δεχτούμε. Λοιπόν, εξαρτάται, ε, ε, δεν νομίζω ότι αυτή ήταν ε, η πρόταση του νομοθέτη που συνέταξε τις συνθήκες. δεν ήθελε προφανώς να δημιουργεί τέτοιες αμφίσιμες καταστάσεις όπου δύο θεσμικά όργανα τσακώνονται για το του πιουνού ε, οργάνου η πρόταση θα υπερισχύσει. Και γι' αυτό ότι ε, όταν θα υπάρξει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νομίζω ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να αφήσει την Επιτροπή να κάνει σωστά τη δουλειά της. Διαφορετικά θα καταλήξουμε σε πολλά προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σντάνοκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βαρόνι Λάτφορτ για τη θαυμάσια δουλειά της. Ε, είμαι πεπισμένη ότι προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μιλήσω εκ μέρους των βουλευτών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ελεύθερη, στον Ευρωπαϊκό Ελεύθερο Συνασπισμό που εκπροσωπεί τις μειονότητες και τις μη επίσημες ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι η διερμηνία και η μετάφραση των εγγράφων θα πρέπει να εξασφαλίζεται και στις μειωτικές γλώσσες. Παραδείγματο χάρη, σε εκείνες τις δικαιοδοσίες όπου χρησιμοποιούνται αυτές οι μειωνοτικές γλώσσες και θα, θα πρέπει τότε να υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γλώσσες. Είναι κρίμα που η Ευρωπα... ο Ευρωπαϊκής Χάρτης για τις περιφερειακές και μειωνοτικές γλώσσες δεν είναι τμήμα του κοινωτικού κεκτημένου. Είμαι σίγουρη όμω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα συμβεί αυτό και η χρήση αυτών των γλωσσών στι ποινικέ ε, διαδικασίε θα εξασφαλιστεί ε, και θα κατοχυρωθεί και μέσω και του ευρωπαϊκού δικαίου. Η κυρία Γκάλ για δύο λεπτά. Κυρία Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια για την ε, συνεχή προσπάθειά της. Εδώ και χρόνια διαπραγματευόμαστε αυτό το πακέτο και χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας τελικά αυτές οι διατάξεις ε, μετά την απόφαση του Συμβουλίου ειδικά θα εφαρμοστούν. Αυτή η οδηγία είναι πάρα πολύ σημαντική, θεμελιώδης, γιατί τη μέρα που, σε μια εποχή που μπορούμε να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, όταν ένας πολίτης αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση όπως είναι μια ποινική διαδικασία, καλό είναι να τον καταλαβαίνουν και να καταλαβαίνει τι του λένε. Μετά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και την πρωτοβουλία που ανελήφθη, θα έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και σε αυτό το τομέα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ακριβώς μας επιτρέπει να προχωρήσουμε προς το συμφέρον των πολιτών μας η σημασία της Ευρωπαϊκής Χάρτας που θα ενσωματωθούν μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και τη σύμβαση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει αλλά θα γίνει. Θα ήθελα να συμπαθυμίσω κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Οι πολίτες που ανήκουν σε μειονότητε, κανονικά θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα στα πλαίσια μιας ποινική δίκης με τους πολίτες που βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Επομένως, θα πρέπει χάρη στην νομοθεσία ο καθένας να μπορεί να χρησιμοποιεί την ε, μητρική του γλώσσα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτή την αρχή ε, σε περίπτωση που ένας πολίτης χρησιμοποιεί μια μειονοτική γλώσσα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να είναι υποχρέωση των κρατών μελών. Ο κύριος Κοέγιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν κατέληξαν σε συμφωνία και τελικά μπλοκάρισαν την πρώτη απόπειρα για ένα ε, νομικό μηχανισμό που θα δώσει ε, μεγαλύτερη ομοιογένεια στις διάφορες οικονομικές διαδικασίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. τώρα αντικαθίσταται από μια, μια προσπάθεια πρόοδου. Έξι μέτρα λοιπόν στην προσπάθεια τη δεύτερη για τη γραπτή μετάφραση, κάτι το οποίο δεν υφίσταται ακόμη σε όλα τα κράτη-μέλη και όταν υφίσταται ως δικαίωμα υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Δικαίωμα διερμηνίας, κάτι το ούτε αυτό είναι κατοχυρωμένο. Όλοι λοιπόν οι ύποπτοι κατηγορούμενοι θα έχουν τη νομική συνδρομή πλέον μέχρι το τέλος, μέχρι το πέρας της δίκης. Έτσι ανταποκρινόμαστε ε, στις μείζονες ανησυχίες του Κοινοβουλίου μετά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλω να συγχαρώ την κυρία Ρέντινγκ, η οποία έχει υποβάλει μια πολύ καλή πρόταση. Θέλω να συγχαρώ και την κυρία Λάντφορντ, διότι κατέληξε σε ένα συμβιβασμό για όλα τα σημεία και δει τη γραπτή μετάφραση των βασικών στοιχείων των δικογράφων έτσι ώστε το επίπεδο να μην είναι ποτέ χαμηλότερο αυτού που προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Χάρτα. Τώρα θα πρέπει βέβαια να δούμε ε, κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα προχωρήσουν σε ταχεία εφαρμογή και δεν θα αφήσουν για την τελευταία στιγμή την ε, μετάταξη στο εθνικό δίκαιο αυτού του ε, νομικού κειμένου. Κυρία Ρέντινγκ, ελπίζω να μπορέσετε να μας υποβάλλετε ως συνέχεια ε, αυτή τη απόπειρα και άλλες προτάσεις, είναι προφανέ ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη δικαιοσύνης και όχι μόνο μια Ευρώπη ελευθερίας και ασφάλειας. Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι όλες οι χώρες πλήν τη Δανία συμφωνούν να τηρήσουν τα πρότυπα αυτά και η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν να ασκήσουν επίση το δικαίωμα του opt-in. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, στα πλαίσια του Catch the ο κύριος Βος είναι ο πρώτος μιλητής. Ευχαριστώ, <clears throat> κυρία Επίτροπε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι ε, τόσο πολύ μάχεστε ε, για τα διαδικαστικά δικαιώματα όσον αφορά στις δίκες και είμαι πολύ ευτυχής που καταφέραμε χάρη στην κυρία Αντωνέσκου να αφαιρέσουμε τα επουσιώδη θέματα από την έκθεση αυτή. Καλό θα ήταν να ζητήσουμε περισσότερα από τους μεταφραστές. Δηλαδή θα πρέπει κανείς να έχει εξασφαλίσει την ποιότητα της μετάφρασης. Η τα τρία χρόνια ίσως ε, είναι πόδινα αλλά δευτερεύον θέμα ουσιαστικά και ε, θα καταλήξουμε στο σεβασμό της ε, συνθήκης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε μη ευθυγράμμιση των νομομαθών οπότε σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις κινήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η έκθεση αυτή είναι μία πρόεδρος για την Ευρώπη. Είναι πολύ, ένα πολύ καλό βήμα για να υπάρξει μία Ευρώπη δικαίου. Πολλά όμως θα εξαρτηθούν από την ενιαία εφαρμογή που είναι απαραίτητη διότι μόνο τότε ε, θα μπορέσει κανείς να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Εγώ θα ήμουν πολύ ικανοποιημένη αν μπορούσε κανείς να λύσει και τα θέματα των διαδικαστικών ποινών διότι πολλά από τα θέματα δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το μέτρο αλλά το πεδίο είναι πολύ ευ ευρύ και ελπίζω ότι σε εφαρμογή του προγράμματος της Σοκχόρμης θα καλυφθούν και τα υπόλοιπα θέματα. Ευχαριστώ κύριος Μπάτεν. Το βασικό πρόβλημα με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα δεν είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, διερμηνία, αλλά είναι ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι αδύναμα για να προστατεύσουν τους υπηκόους του εναντίον ε, των άδικων εκδόσεων. Ο άντιο Σίμιο από την εκλογική μου περιφέρεια κρατήθηκε 11 μήνες σε μια ελληνική φυλακή στον Κορυδαλό, περιμένοντας τη δίκη. Διάφοροι άλλοι πολίτες, έξι πολίτες, ε, αντιμετωπίζουν το φάσμα της ε, έκδοσης και παραμένουν στο Κορυδαλό. Και οι Βρετανικές αρχές δεν μπορούν να εξετάσουν ε, τις, τα στοιχεία που υπάρχουν αντίον τους. Ε, στον Κορυδαλό, ε, πάρα πολύ φυλακισμένοι, ε, περισσότεροι από ό,τι πρέπει βρίσκονται στο ίδιο κελί. Υπάρχει βία, οι τουαλέτες είναι και ακούγονται φωνές το βράδυ. Η, Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να ντρέπεται που χάρη μέσω ένα... ενός χαρτιού εκχωρεί δικαιώματα των Βρετανών υπηκόων υπέρ ενός μέρους που είναι πραγματικά αηδέ. Thank Ευχαριστώ. Είναι προφανώ ε, σωστό ότι όσοι βρίσκονται σε οικοδομικέ διαδικασίε θα πρέπει να έχουν υπηρεσίε μετάφραση και διερμηνία, ιδίω εφόσον το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη ε, προβλέπει έκδοση ατόμων για ε, δικήματα που δεν είναι δικήματα στη χώρα καταγωγή του. Ωστόσο, αυτό είναι ένα από τα μη από τα λεγόμενα τιμήματα του εντάλματος όταν αυτό προτιοθετήθηκε. Παπα-Νικολάου. Παπα νικολαου θελω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ γόνιμη συνεργασία που είχαμε. Πολλοί από εμά στην Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιοσύνη υποβάλαμε τροπολογίε σε αυτή την έκθεση, την τόσο σημαντική έκθεση, και συμπεριλαμβάνονται πλέον στο τελικό κείμενο. Πράγματι η διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ε, είναι γόνιμα τα συμπεράσματα και πράγματι καταλήγοντας και φτάνοντα στο σημείο τη ψήφιση αυτή τη οδηγία οφείλουμε όλοι να αναγνωρίσουμε ότι στα πλαίσια των ποινικών διαδικασιών θεμελιώνουμε ακόμη περισσότερο την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των αλλόγλωσσων κατηγορουμένων. έχει πολύ μεγάλη όμως σημασία κυρία επίτροπε επειδή και η τριετία που θα έχουμε μπροστά μας στα πλαίσια αυτού του οδικού χάρτη για την εφαρμογή είναι αρκετός χρόνος περιμένουμε πολλά από την επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και τα χειροπιαστά αποτελέσματα μετά την ενσωμάτωση αυτής τη οδηγία. Ε, έχουμε μεγάλες προσδοκίες ευελπιστούμε ότι θα αλλάξουν πολλά έχει σημασία όμω να μην τα αφήσουμε όπω πολύ σωστά υπόθηκε και από τους συναδέλφους προηγουμένως ε, να μην τα αφήσουμε όλα για την τελευταία στιγμή. Σα ευχαριστώ πολύ. Η θα απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές οι οποίοι με ένα πολύ πιστικό και στεναρό τρόπο υποστήριξαν τον τομέα της δικαιοσύνης που έχουμε αρχίσει να οικοδομούμε. Το χώρο της δικαιοσύνης που έχουμε αρχίσει να οικοδομούμε. Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει, μας δίνει τώρα την ευκαιρία, γιατί μας δίνει τα κατάλληλα εργαλεία, να προχωρήσουμε βαθμιδών για να δημιουργήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Που σημαίνει δικαιώματα και θυμάτων και δικαιώματα και των καταδίκων. Τώρα, περισσότερες προτάσεις στα πλαίσια του οδικού χάρτη θα υπάρξουν. Αυτό ήταν μια ερώτηση. Ναι, Πρόεδρε. Μετά το δικαίωμα στη διερμηνία, που είμαι σίγουρη ότι θα υποψηφίσετε αύριο, θα υπάρχει το δικαίωμα στην ενημέρωση. Η επιστολή των δικαιωμάτων που θα υποβάλω ε, στους βουλευτές πριν από το καλοκαίρι. Εν συνεχεία, θα έχουμε το δικαίωμα σε νομική συμβουλή και το δικαίωμα σε επικοινωνία με τους αγαπημένους σου. Πηγαίνουμε λοιπόν προς μια κατεύθυνση η οποία θα μας επιτρέψει να, επιτύχουμε τα εξής. Να έχουμε τα ίδια δικαιώματα σε ένα υψηλότατο επίπεδο για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και αν βρίσκονται. Όποιο και είναι το πρόβλημά τους, είτε ταξιδεύουν για σπουδές, για τη δουλειά τους ή για ψυχογεία, δεν έχει καμία σημασία. Δεν, πρέ... έχει σημασία αυτό. Θα πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους και να έχουν τα ίδια δικαιώματα με την πατρίδα τους, όπου και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Τώρα, μία σημαντική ερώτηση, την οποία επανέλαβαν πολλοί βουλευτές. Το θέμα της γλώσσας και των γλωσσών εν γέννη. Αν κοιτάξω το άρθρο 2, εδάφιο 1 και το άρθρο 3 εδάφιο 1, λέγεται ξεκάθαρα ότι ο κατηγορούμενος ο οποίος δεν καταλαβαίνει ή δεν μιλάει τη γλώσσα του δικαστηρίου θα πρέπει να έχει ένα διερμηνέα. Και επίσης θα πρέπει να του μεταφράζονται τα έγγραφα. Αυτό έμεσα σημαίνει ότι η γλώσσα στην οποία του μεταφράζονται τα έγγραφα είναι μια γλώσσα την οποία καταλαβαίνει. Ακόμα δεν περιοριζόμαστε στις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε καν στις μειονοτικές γλώσσες. Μιλάμε για τη γλώσσα του εκάστοτε ανθρώπου που βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου και αντιμετωπίζει κατηγορίες. Νομίζουμε ότι αυτό είναι δίκαιο, γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη δίκη για όλους ούτως ώστε να υπάρξει εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα δικαιοσύνης. ούτως ώστε να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη των, και των δικαστών και των εισαγγελέων στα συστήματα των γειτονικών χωρών. Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο αν έχουμε το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων. Μία άλλη ερώτηση ακούστηκε από τον κύριο Μπουσουτήλ και από άλλους βουλευτές. Όχι για τα δικονομικά δικαιώματα, αλλά για τις εσωτερικές διαδικασίες. Γιατί συνυπάρχει μία πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους και η πρόταση της Κομισιόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα η, να υιοθετηθούν γρήγορα και με ισορροπημένο τρόπο ε, νομοθετικά εργαλεία. Γιατί έχουμε αυτές τις παράλληλες πρωτοβουλίες. Βρισκόμαστε σε μια ιδιάζουσα περίοδο. Βγαίνουμε από τον τρίτο πυλώνα και μπαίνουμε σε μια συνήθη διαδικασία συναπόφασης. Υποθέτω ότι μετά από κάποιους μήνες θα έχουμε μάθει πώς θα χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ούτω ώστε πολύ γρήγορα να βρίσκουμε την καλύτερη λύση. Και όταν μιλάω για την καλύτερη λύση, ενώ όπως ακριβώς ετοιμάζαμε αυτές τις ε, λύσεις, κάνοντας μία μελέτη αντικτύπου, υποβάλλοντας προτάσεις, ούτως ώστε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον ε, για να μας πει ο κόσμος τι πιστεύει για τις ε, προτάσεις μας. Τι συνήθειες διαδικασίες που χρησιμοποιούσαμε και που στο τέλος, μέσω της διαδικασίας της συναπόφασης και μετά από μια δημόσια διαβούλευση και μετά από τη μελέτη αντικτύπου, εξασφαλίζουν ότι προβαίνουμε σε υγιείς και σωστές πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες εν συνεχεία να μπορούν να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο χωρίς στρεβλώσεις και χωρίς προβλήματα. Κάτι που δυστυχώς ε, έχει συμβεί στο παρελθόν. Σήμερα είμαστε εδώ με μια νέα συνθήκη. Έχουμε τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, θα γίνουμε συμβαλόμενο μέρος της ε, Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χάρη σε αυτό είμαι πεπισμένη, σε όλα αυτά είμαι πεπισμένη ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα, όταν ξανασυναντηθούμε, θα διαπιστώσουμε με ικανοποίηση ότι οικοδομήσαμε μαζί αυτό το χώρο δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων για την Ήπειρό μας. Ευχαριστώ την Επίτροπο. Και τώρα η Βαρόνη Λάτφορντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ειλικρινέστατα να ευχαριστήσω τους ποιοτικότατους οδησυχητές για τη βοήθειά τους. Χαίρομαι που συζητούμε και ψηφίζουμε επί Ισπανικής Προεδρίας αυτή την έκθεση. Πρόκειται για ένα ιστορικό μέτρο, το πρώτο μέτρο που συζητούμε στο πλαίσιο της διαδικασίας εναπόφασης και συμφωνώ και με τον Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ για την τριετή περίοδο εφαρμογής. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ε, ακαθόδες το θέμα ε, μετά την συμφωνία. Κάποιοι προσπάθησαν μονομερό κάποια κράτη-μέλη να κάνουν τα δικά του, δεν θα του περάσει όμω τώρα. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε, να ακολουθούμε εθνικιστικέ ε, προσεγγίσεις για αυτά τα ζητήματα. Στρέφομαι στον ανθρώπου από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις ε, με τις 20 μέρες κάθριξης ε, χωρίς απαγγελία κατηγορία κτλ. Και ελπίζω μια κυβέρνηση να αλλάξει κάποια πράγματα. Η οδηγία πάντως αυτή θα καλύπτει 26 χώρες και διαπνέεται από το πνεύμα του Χάμπιου Κόρπου τη Μάγνα Κάρτα και του, δικαιο... του νομοσχεδίου του νόμου για τα δικαιώματα, του Bill of Rights, ώστε οι ε, παρανομούντες να μην ε, διαφεύγουν τη δικαιοσύνη Ό,τι αφορά ε, το δικαίωμα χρήση περιφερειακών μειονοτικών γλωσσών. Συμφωνώ με τις τροπολογίε που μάλλον τις κατανοώ, αλλά δεν μπορώ να τι δεχθώ. Διότι ο στόχο είναι η συνεκτικότητα, η συνεπικανότητα να μιλά κάποιο, να εκφράζεται ε, και ε, όχι να επιλέγει τη γλώσσα που θέλει. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει μια διαδικασία παλήθευση τη ικανότητα ενό ατόμου να καταλαβαίνει ή να μιλά τη γλώσσα. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε μπορεί να υπάρξει αποσβολή μια απόφαση. Σε ό,τι αφορά τα μειονοτικά δικαιώματα, πρέπει να πω ότι αυξάνονται στην πράξη τα δικαιώματα αυτά στο βαθμό που ο μιλητή μια μενοτική γλώσσα που δεν μπορεί να καταλάβει ε, τη διαδικασία, ε, σε αυτόν ισχύουν ε, τα δικαιώματα τα οποία προβλέπει η οδηγία. Ελπίζουμε λοιπόν να περάσει χωρίς τροπολογίες και γρήγορα και στο καταστατικό αυτή η τροπολογία και η, μάλλον αυτή η πρόταση και ελπίζω να έχουμε σύντομα τα πρώτα μέτρα. μέσα σε 15 μέρες είναι τα πρώτα και στα χέρια άλλωστε της πάρα πολύ μαχητικής αντιπροέδρου μας νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε προκαλέσει ερώτημα από τον κύριο Μπάτεν, κύριε Λάτφορντ. Το δεχθείτε, ναι. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Μπάτεν. Ευχαριστώ πολύ, Βαρόνι Λάτφορντ. Έχετε ξαναπεί στο παρελθόν συζητήσει αυτές ότι εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των γκάγκστερ στην Κώστα Σόλ. Κάτι αντίστοιχο είπατε και σήμερα. Έχετε ένα στοιχείο όμω για τον αριθμό των εγκληματιών, των, ε, κλεπτών, των διαρρηκτών τραπεζών ε, που έχουν συλληφθεί από την Κώστα Ντελσόλ αφότου άρχισαν να ισχύει το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη. Όχι. Όχι, θα το ψάξω, κύριε Μπάτον, και θα σα ενημερώσω για το νούμερο. Και εγώ να σα ρωτήσω κάτι με την ε, σειρά μου. Ε, και, εγώ και εσείς εκπροσωπούμε το Λονδίνο. Ε, το Ιούλιο του 2005 ένας βομβιστής ε, διέφυγε προς την Ιταλία. Ελπίζοντας, φαντάζομαι, ότι θα εξαφανιστεί εκεί. Στο παρελθόν θα μπορούσε να κρύβεται για χρόνια. Εδώ τον, μας τον επέστρεψαν μέσα σε έξι εβδομάδες και τώρα καταδικάστηκε και με βάση τον νόμο και την τρομοκρατία ε, εκτεί την ποινή του. Φαντάζομαι θα θέλατε να μην είχε δικαστεί ποτέ. Αυτό θα θέλατε. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, έκλεισε η συζήτηση τώρα. Και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη. Και τώρα πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση Κλούνα για την υιοθέτηση από την